Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Θα αρχίσουμε με ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την σύμβαση για τον ε, κυβερνοχώρο και τα κλίματα στον κυβερνοχώρο με το Συμβούλιο. Ξέρετε ότι εξετάζουμε αυτό το θέμα εδώ και καιρό. Πολλοί από εσά είσαστε αρκετά ειδικοί και για τους νέους ευρωβουλευτές, όπως μας δήλωσαν, είναι ζωτική σημασία η έρευνα που γίνεται γι' αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι και το Μάρτιο που μας πέρασε εκδηλώσαμε την ανησυχία μας όσον αφορά την τακτική και το πώς προχωράει με τα διάφορα άρθρα η ομάδα εργασίας που ασχολείται με την σύμβαση αυτή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό θέμα για μας και σας παρακαλώ να ασχοληθείτε όλοι γιατί σίγουρα θα δουλέψουμε πολύ πάνω σε αυτό το θέμα μέσα στους επόμενους μήνες. Έχει μεγάλη σημασία η καταπολέμηση του κλίματος στον κυβερνό Ξέρω ότι ορισμένοι συμμετέχουν στην έρευνα και εννοείται ότι θα τους ακούμε τακτικά. Ας περάσουμε στις παρουσιάσεις. Έχουμε εδώ τους προσκεκλημένους μας. Καλώς ήρθατε όλοι. Πρώτα απ' όλα έχουμε τον Αλεξάνδερ Σίκερ, ο οποίος είναι εκτελεστικός γραμματέας της Επιτροπής της Σύμβασης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. ΣΥΠΡΟΚ. Εδώ θα υπάρξει πολλή ορολογία σήμερα. ΣΥΠΡΟΚ. Και μετά έχουμε τον Eric Plankton που είναι από το CTI. Μπορείτε να μας εξηγήσετε εσείς περί τίνος πρόκειται, τι ακριβώς είναι αυτό. Τι είναι το ΣΥΠΡΟΚ, κύριε Πλάνκεν. Τον Τζοβάνι Μπουταρέλη θα το ξέρετε γιατί είναι ο αναπληρωτής ε, του, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Και έχουμε και τον Βότσκες Ράφαλ Βιβιόροφσκι που είναι γενικός επιθεωρητής για την προστασία των δεδομένων. Είναι στην ομάδα εργασίας του άρθρου 29. Θα το ξέρετε. Είναι αντιπρόεδρος αυτή την ομάδα εργασίας. Συνεπώς, αγαπητοί συνάδελφοι, θα μοιράσετε μεταξύ σας το χρόνο και τις παρουσιάσεις. Έρικ, θα ακούσουμε σένα πρώτα. Και μετά οι ευρωβουλευτές θα υποβάλουν ερωτήσεις. Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Ως πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής που ασχολούνται με τη σύμβαση της Βουδαπέστης, το TCY, όπως είναι τα αρχικά, θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω για το έργο της Επιτροπής μας και να σας πω τι κάνουμε για την προστασία των δεδομένων. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σύνθετο θέμα. Γι' αυτό θα παραμείνω αρκετά γενικό στα σχόλιά μου, επειδή έχουμε περιορισμένο χρόνο. Καταρχήν, ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής μας ρυθμίζεται από άρθρο 46 της Σύμβασης για να διασφαλίσει την ίδια τη λειτουργία της Σύμβασης. Πρώτα απ' όλα αξιολογεί την εφαρμογή από τα διάφορα μέρη. Δηλαδή αυτή την εποχή εξετάζουμε πόσο αποτελεσματικές είναι οι διατάξεις για την νομική αρρωγή από την σύμβαση αυτή βάσει αρετηματολογίων και συζητήσεων που κάνουμε στην Επιτροπή μας. Δεύτερος ρόλος μας είναι να εκδίδουμε κατευθυντήριες γραμμές για τις διατάξεις της σύμβασης για να δούμε πώς μπορούν να εφαρμόζονται πιο αποτελεσματικά εξετάζοντας φαινόμενα τα οποία ίσως δεν υπήρχαν όταν καταλήξαμε στην ε, σύμβαση αυτή. Για παράδειγμα, είχαμε κατευθυντήριες γραμμές για το να ασχοληθούμε με θέματα κλοπής ε, ταυτοτήτων ή ε, αλλά τα οποία ίσως παλιότερα να μην είχαν την ίδια σημασία. Τρίτος ρόλος μας είναι να ετοιμάζουμε νέα πρωτόκολλα στη σύμβαση αυτή. Εξετάζουμε δηλαδή πόσο εφικτό είναι να προσθέτουμε ένα επιπλέον πρωτόκολλο για θέματα προστασίας δεδομένων. Υπογραμμίζω εδώ ότι η σύμβαση της Βουδαπέστης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι κάτι που έχει να κάνει ακριβώς με το έγκλημα και μερικές φορές αυτό δεν γίνεται κατανοητό. Η σύμβαση απαιτεί δηλαδή να αποφασίσουν για το εγκληματικό χαρακτήρα διαφόρων παραπτωμάτων οι χώρες μέλη και ζητάει από τα διάφορα μέρη να φροντίζουν να έχουν τις εξουσίες ώστε να συγκεντρώνουν ηλεκτρονικά στοιχεία για οποιοδήποτε έγκλημα και ζητά επίσης από τα διάφορα μέρη αποτελεσματικά να συνεργάζονται μεταξύ τους και σε διεθνές επίπεδο. Στόχος ε, λοιπόν είναι το άρθρο 40 και οι εξουσίες που προσφέρουν οι συνθήκες και να εφαρμόζονται σε δεδομένα που περνάνε σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε σχέση με κλιματικές πράξεις. Το άρθρο 50 λέει ότι οι εξουσίες αυτές πρέπει βέβαια να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δίκαιο. Και για να είμαστε σαφείς εδώ, ετοιμάζοντας μια κατευθυντήρια γραμμή για παράδειγμα, ή όταν σκεφτόμαστε αν πρέπει να προσθεθεί πρωτόκολλο, στόχος μας δεν είναι να επεκτείνουμε το εύρος ε, της σύμβασης αυτής, να καλύψουμε δηλαδή παραπάνω θέματα, όχι. Το θέμα της πρόσβασης σε δεδομένα στα πλαίσια εγκληματικών πράξεων, ερευνών για εγκληματικές πράξεις, καταλαβαίνετε ότι διαφέρει πολύ από το θέμα της ε, μαζικής εποπτείας που αναλαμβάνουν εθνικοί οργανισμοί ασφάλειας. Εδώ και πάλι πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι καθόλου πρόθεσή μας να προσθέσουμε επιπλέον στοιχεία ή να παρέμβουμε σε άλλες δικαιοδοσίες όπως έχουμε δηλώσει πρόσφατα. Το έργο μας λοιπόν για την πρόσβαση σε δεδομένα γίνεται για τον εξή λόγο. Γιατί πολλέ φορέ τα δεδομένα σε ε, δικαστικέ ε, διαδικασίε αποτελούν ε, αποδεικτικά στοιχεία και πρέπει να υπάρχουν χωρί καθυστέρηση. Γι' αυτό και έχουμε συμπεριλάβει στη Σύμβαση τη Βουδαπέστη διάφορε ειδικέ αρμοδιότητε που όμως εφαρμόζονται σε πολύ περιορισμένε περιπτώσει. Το άρθρο δεν επαρκεί είναι από το 2001. Ούτε ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τις πληροφορίες ο κόσμος είναι ίδιος όπως ήταν τότε, καθόλου. Δύσκολα βέβαια μπορεί κανείς να καταλήξει σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Υπάρχει και το cloud. Οι αρχές, οι δικαστικές που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό έγκλημα ε, βέβαια έχουν ένα πολύ δύσκολο ρόλο αλλά και για άλλους λόγους, είτε οικονομικούς είτε άλλους, τα δεδομένα πολλές φορές φεύγουν, εξαφανίζονται, πηγαίνουν αλλού και είναι δύσκολο να εντοπιστεί το σημείο από όπου έχουμε τα δεδομένα αυτά. Γι' αυτό και χρειάζεται αμοιβαία αρρωγή για να μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο όπου βρίσκονται τα δεδομένα και πρέπει να ξέρουμε, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 32 για παράδειγμα, πού πρέπει να στραφούμε. Το ηλεκτρονικό έγκλημα αυξάνει εκθετικά με το διαδίκτυο βέβαια, αλλά όχι μόνο. Ξέρετε ότι κανείς ε, μπορεί, άμα θέλει, ακόμα και όπλα και ναρκωτικά ή να παραγγείλει μια δολοφονία ή έναν βιασμό με το λεγόμενο βαθύ διαδίκτυο. Αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών που έχουμε τα τελευταία χρόνια, οι δικαστικές αρχές είναι όλο και λιγότερο σε θέση να προστατεύσουν την κοινωνία και τα άτομα από το έγκλημα. Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών, μάλιστα, δεν είναι δυνατόν καν να γίνουν γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση σε δεδομένα και έτσι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο σε πολλές περιπτώσεις μένει ατιμόρυτο. Και αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνο με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Και αυτό δεν είναι αλήθεια μόνο για μικρά παραπτώματα, αλλά και για άλλε περιπτώσεις βίας ή πολύ άγριων εγκλημάτων. Τα θύματα και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους πολλές φορές παραβιάζονται. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Η δικαιοσύνη όμως δεν είναι δυνατόν να είναι ελλειπής επειδή δεν υπάρχουν ε, δεδομένα. Οι κυβερνήσεις λοιπόν είτε έχουν ήδη κάνει ρυθμίσεις για διμερείς ή μονομερείς ε, λύσεις προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα. Ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου να μην μπορούν να βρεθούν λύσεις. Όταν όμως λύσει. λύσεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό όμω μονομερό η διμερο βρισκονται λύσει, μάλλον η Επιτροπή, θέλει να οδηγησει σε ζουγκλα Όπω ειπα και νωριτερα η συμβαση η μαλλον η επιτροπη θελει να αντιμετωπισει τι προκλήσει αυτέ και το 2011 αποφασίσαμε να δούμε τι δυνατότητες έχουμε, τι παραπάνω δυνατότητες έχουμε για να διευκρινιστεί το άρθρο 32β και στα μέσα του 2013 ετοιμάσαμε σημειώματα με κατευθυντήριες γραμμές και το Δεκέμβριο του 2013 τα συζητήσαμε. Όμως δεν προχωρήσαμε ακόμα γιατί, όπως συγκεκριμένα αναφέρεται, χρειάζεται περισσότερο διάλογος με τις αρχές προστασίας δεδομένων, τον Ευρωπαίων Πόπτων Δεδομένων δηλαδή και την κοινωνία των πολιτών ώστε να υπάρχουν αρκετές ρήτρε διασφάλισης και προστασίας των ατόμων και να μην γίνονται καταχρήσεις. Έπειτα είπαμε ότι ενώ η σύμβαση της ε, Βουδαπέστης είναι μια συνθήκη για την καταπολέμηση του κλίματος στον κυβερνοχώρο, υπάρχουν εκθέσεις από διάφορα Ινστιτούτα Εθνικά για την Ασφάλεια που επηρεάζουν τελικά το εύρος εφαρμογής της σύμβασης αυτής. Όπως σας είπα, λοιπόν, αξιολογούμε και το θέμα της αμοιβαία νομικής αρρωγής και της συνεργασίας, κάτι το οποίο θα οδηγήσει πολύ πιθανόν σε επιπλέον προτάσεις για νέο πρωτόκολλο. Προκειμένου τώρα να έχουμε περισσότερο διάλογο, είχαμε μια δημόσια κρόαση τον Ιούνιο του 2013 με ομάδες εργασίας επίσης και με ολομέλειες το 2013. Φέτος το Μάιο είχαμε μάλιστα μια συνάντηση με εκπροσώπους της Ομάδας Εργασίας 29, τον Επόπτη Προσωπικών Δεδομένων και τη Συμβουλευτική Επιτροπή της Σύμβασης για την Προστασία Δεδομένων 108. Και τον Ιούνιο που μας πέρασε είχαμε και μια διάσκεψη για την επιβολή του νόμου και πρόσβαση σε δεδομένα. Η Επιτροπή για τη Σύμβαση που αντιμετωπίζει το έγκλημα στον, το, στον κυβερνοχώρο έχει βέβαια πολύ δύσκολη δουλειά. Χρειάζεται τη συνεργασία όλων των πλευρών. Μερικές φορές υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις όταν βιαζόμαστε στο να υποβάλουμε μία πρόταση. Και η περίπτωση του 32 είναι μία τέτοια. Κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχουν απλές λύσεις. Πιστεύουμε όμως ότι πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο. Το Δεκέμβριο έχουμε την επόμενη ολομέλειά μας, η οποία θα ασχοληθεί με το πώς θα συνεχίσουμε. Όπως έχουν τώρα τα πράγματα, δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση, εξετάσουμε το ενδεχόμενο νέο πρωτοκόλλου μόνο για το περιεχόμενο του σημείου 32. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εκτελεστικό γραμματέα της Επιτροπής μας τον κύριο Αλεξάνδερ ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να προσθέσω έξι σημεία και έχω και κάποια ερωτήματα που θέλω να θέσω. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την ακρόαση. Χρειάζεται να ανταλλάσσουμε πιο συχνά απόψεις, όχι μόνο ε, μεταξύ της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και της Επιτροπής ε, για το κυβερνό έγκλημα. Αλλά να πω ότι και η Εστονία στο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι υπεύθυνη για αυτά τα ζητήματα και μας ενδιαφέρει με μια πιο δομημένη συνεργασία με την Επιτροπή, την Επιτροπή σας. Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Σεπτεμβρίου του 2013 αναφέρεται η συνθήκη της Βουδαπέστης γιατί ε, χρειάζεται μια τέτοια στρατηγική καθώς ε, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι πολύ καλή η προσπάθεια του Συμβουλίου της Ευρώπης να ανανεώσει τη σύμβαση έτσι ώστε να αντιμετωπίσει το έγκλημα στον κυβερνό χώρο. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Η επικοδομητική συνεργασία λοιπόν είναι απαραίτητη για να βρεθούν οι αποδεκτές λύσεις. Οι απόλυτες δηλώσεις και θέσεις δεν είναι επιθυμητές. Τέταρτον, η Επιτροπή για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο ήταν διαφανής και μπήκε σε διάλογο από την αρχή. Γιατί κάθε λύση πρέπει να συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Και όπως αναφέρεται ήδη σε διάφορες ε, συναντήσεις και ανταλλαγές απόψεων που είχαμε με διάφορα μέρη και ενδιαφερόμενους φορείς και πραγματικά κάθε τρεις μήνες υπάρχει μια συνάντηση με διαφορετική σύνθεση ε, αυτό που πάντοτε προκύπτει είναι ότι πρώτον ε, υπάρχει θέμα ε, η ποινική δικαιοσύνη έναντι της εθνικής ασφάλειας. Η σύμβαση της Βουδαπέστης έχει να κάνει με την ποινική δικαιοσύνη, έχει να κάνει με τις ανακριτικές διαδικασίες για συγκεκριμένα δεδομένα. Επίσης, χρειάζεται ένας εθνικός διάλογος για θέματα εθνικής ασφάλειας και ποινική διαδικασίας. Γι' αυτό χρειάζεται καλύτερη εποπτεία, ρύθμιση και έλεγχος των εθνικών διατάξεων για την εθνική ασφάλεια. Των διατάξεων για την εθνική ασφάλεια. Επίσης υπάρχει ένα πλαίσιο που εφαρμόζεται για την προστασία των δεδομένων. Στο επίπεδο της ποινική δικαιοσύνης ε, αλλάζουν τα πλαίσια και γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια πιο σφαιρική άποψη ε, ούτε το Συμβουλίο της Ευρώπης, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, μόνοι τους ε, απομονωμένοι. Υπάρχουν πάρα πολλά κράτη που δεν είναι μέλη μας και δεν θα πρέπει να υπάρχει αντίφαση μεταξύ της Σύμβασης της Βουδαπέστης και της Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και οι δύο προστατεύουν τα άτομα από επιθέσεις προς την ιδιωτική του ζωή η συνθήκη της Βουδαπέστης θέλει να προστατεύσει την ακεραιότητα, την ε, διαθεσιμότητα και την εμπιστευτικότητα των ε, ε, δεδομένων. Αυτές οι δικλείδες ασφαλείας λοιπόν είναι το πιο δύσκολο σημείο. Στο στάνταρ σενάριο όμως, όταν ένας ύποπτος υπόκειται σε μία νόμιμη διερεύνηση και τα δεδομένα του είναι στο εξωτερικό, γιατί να μην εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους που διερευνά την υπόθεση. Επίσης μπορεί να δίνεται δυνατότητα ηθελημένης και κούρσιας αποκάλυψης των δεδομένων. Το άρθρο 29 και πολλά άρα σχετίζονται με αυτό. Να μπορούν δηλαδή οι παροχές υπηρεσιών ε, εθελούσια να αποκαλύπτουν πληροφορίες. Και το άρθρο 32 επίσης λέει για αυτούς ότι δεν θα μπορούν μάλλον να συνενέσουν σύμφωνα με το άρθρο 32 ε, στην αποκάλυψη αυτών των δεδομένων. Παρ' όλα αυτά δεν γνωρίζουμε αν αυτό ισχύει ως ε, δήλωση γιατί υπάρχουν πιθανότητες υπαρχής υπηρεσιών να μπορούν να αποκαλύψουν εκούσια τα δεδομένα. Κάτι άλλο που έχει προκύψει από τις ε, συζητήσεις είναι ε, αν θα πρέπει να ρυθμίσουμε ή να αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν μόνα τους. Θα πρέπει να βάλουμε ένα πρωτόκολλο στην σύμβαση της ε, Βουδαπέστης ή θα φτάσουμε σε ένα σενάριο ζούγκλας με μια πλειάδα μονομερών διακανονισμών. Αυτά τα θέματα και τα ζητήματα τα θέτω για να αναρωτηθούμε πάνω σε αυτά. Το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των λύσεων είναι πολύπλοκο λοιπόν. Τα πλαίσια προστασίας των δεδομένων δεν έχουν οριστικοποιηθεί ούτε στο Συμβουλίο της Ευρώπης ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκθέσεις για τις μαζικές παρακολουθήσεις ε, μας κάνουν να ανησυχούμε και υπάρχουν πολλά κράτη που παίρνουν επιπλέον μέτρα η απόφαση για την κράτηση των δεδομένων ε, έχει γίνει θέμα πολύ σημαντικό τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει η εξάπλωση του εγκλήματος μαζική, όπως επίσης και των ε, ε, παρεμβάσεων στην ιδιωτική ζωή από εγκληματίες. Και πάλι οι κυβερνήσεις παίρνουν μονομερός λύσεις, μέτρα για να μπορέσουν να λύσουν τα θέματα αυτά. Ε, της πρόσβασης και της μεταφοράς δεδομένων επειδή δεν υπάρχουν διεθνείς ρυθμίσεις. Υπάρχουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις επίσης που αναλαμβάνουν δράση από μόνες τους. Πρόσφατα συναντηθήκαμε με εμπειρογνώμονες ε, που ασχολούνται κυρίως με θέματα της μαύρης οικονομίας και μας είπαν τι δεν μπορούν ε, οι ιδιοκτικές αρχές να βρουν μια IP, μπορούμε να το κάνουμε εμείς, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω λοιπόν να θέσω θέματα στην Επιτροπή, ειδικότερα όσο σχετικά με τα όσα λέει η παράγραφος 32 για το άρθρο 32. Είναι έξυπνη κίνηση να συζητείτε το άρθρο 32 στην παράγραφο 32 της έκθεσης νομίζω. Πώς προέκυψε αυτό, γιατί η Επιτροπή δεν ακούστηκε. Υπάρχει μια σειρά θεσμικών οργάνων που ακούστηκαν από την Επιτροπή σας, γιατί δεν υπήρξε ακρόαση με την Επιτροπή για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο πριν γίνει η έκθεση. Επίσης, η απομακρυσμένη πρόσβαση χωρίς ε, παρεμβάσεις, γιατί να μην είναι δυνατόν να μπορούμε να έχουμε διασφαλίσει σε επίπεδο ποινική δικαιοσύνης, να μην έχουμε εξαιρέσει έτσι ώστε όλα αυτά ε, να θεσπίζουν μια ξεκάθαρη νομική βάση και γιατί η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είναι εναντίον οποιοδήποτε, ε, οποιοδήποτε επιπρόσθετου πρωτοκόλου και πραγματικά προτιμά η Επιτροπή της Μονομερής Λύσης των Κρατών ε, και, των, και τις άτυπες, τους άτυπους διακανονισμούς δεν θέλουν να προστατευτούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των θυμάτων του, ε, των εγκλήματων στον κυβερνοχώρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σαφής η παρουσίασή σας. Ο κύριος Μπουταρέλη στη συνέχεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσά και του συναδέλφου, επειδή καλέσατε τον Ευρωπαίο Πόπτη Προστασία Δεδομένων. Είναι η πρώτη ευκαιρία που είχαμε, που είχαμε να ε, παραστούμε στη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής σας μετά τις εκλογές. Θα χρησιμοποιήσω και τι διαφάνειες αλλά και ε, τα σημεία ομιλίας που σας είχα γνωστοποιήσει. Να σας ενημερώσω καταρχάς τι κάνουμε. Είναι διαθέσιμες οι διαφάνειες. Στα μέσα του 2013 ενημερωθήκαμε για την πρωτοβουλία, για την, ε, πρωτοβουλία ενός επιπλέον πρωτοκόλου και έκτοτε, συγγνώμη κύριε Μπουταρέλη, χρειάζεται διαφάνεια εσάς. Α, είδου. Ωραία. Νάτες. Λοιπόν, μαζί με τους συναδέλφους της ομάδας εργασίας 29, παρακολουθήσαμε τις ε, συζητήσεις, ε, τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο Στρασβούργο. Το επιπλέον πρωτόκολλο σκοπό έχει να αλλάξει άρδιν τις διαδικασίες για την επιβολή του νόμου και τις σχετικές αρχές ε, ως προς την εξαποστάσεως πρόσβαση σε έγγραφα άλλων δικαιοδοσιών. Ε, άλλα θέματα που είναι υποσυζήτηση και τα οποία μπορείτε να τα δείτε τώρα στην παρουσίαση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ο συνάδελφος ε, από την ομάδα εργασίας 29 θα αναφερθεί σε μερικές από αυτές τις επιλογές. Επόμενη διαφάνεια. Στο δικό σας το ψήφισμα του Μαρτίου του τρέχοντος έτους για τα προγράμματα παρακολούθησης ε, γύρατε σοβαρές ανησυχίες γύρω από αυτές τις πρωτοβουλίες και η σημερινή ανταλλαγή απόψεων είναι η συνέχιση του ψηφίσματος αυτού και πρέπει βέβαια να εξετάσουμε τις ανησυχίες που είχατε εκφράσει τότε. Πριν πούμε σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να προσπαθήσω να συνοψίσω κάπως το θέμα. Ο στόχος της τροποποίησης ε, της σύμβασης είναι η διευκόλυνση ε, της ε, ηλεκτρονικής έρευνας που είναι κάτι βέβαια που πρέπει να έχει σχέση πάντοτε με νόμιμους στόχους την πρόληψη και την καταστολή εγκλημάτων. Σε γενικές γραμμές αναγνωρίζουμε την ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας συνεργασίας επιβολής του νόμου και θέλουμε να συνεισφέρουμε προκειμένου να είναι λιγότερο ε, λιγότερο χρονοβόρες. Γνωρίζουμε επίσης η σύμβαση της Βουδαπέστης θέλει να εξασφαλίσει ότι η ε, έρευνες ε, στο πλαίσιο μιας ποινική διαδικασίας ε, δίνουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας να εξασφαλίζεται δηλαδή ότι η πρόσβαση στα δεδομένα από τις αρχές επιβολής του νόμου είναι απαραίτητη και επιλεκτική. Όλες οι εναλλακτικές επιλογές που βρίσκονται υπό συζήτηση αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μας, εξακολουθούν να δημιουργούν πολλές ανησυχίες. Κατά τη γνώμη μας ε, πρέπει να έχουμε μια προσεκτική, μια προσεκτική προσέγγιση ε, πρώτα απ' όλα για τα θε... από εμπιστοσύνης και επίσης ε, υπάρχει και το θέμα της αναλογικότητας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ε, συζήτηση για μια επιλεκτική προσέγγιση. Δεν μπορούμε όμως οι νέες τεχνολογίες να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθούν στο άμεσο μέλλον, πόσο επικίνδυνες και πόσο, πόσο επικίνδυνοι μπορεί να είναι η εξαποστάσεως πρόσβαση. Πρέπει να μην μας διαφεύγει ότι οι διαδικασίες της Σύμβασης Βουδαπέστης ισχύουν για όλα σχεδόν τα εγκλήματα, όχι μόνο για τα εγκλήματα στον κυφέρνο χώρο. Και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ χρήσιμο για τα μέλη της Επιτροπής σας. Βλέπετε πόσο ευρύ είναι το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης. Πρώτον, σε μεγάλη εμβέλεια εγκλημάτων, αυτών που αναφέρονται στην διαφάνεια, αλλά και σε παραπτώματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση υπολογιστών όπως επίσης και με συλλογή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή κάθε ποινικού αδικήματος. Αυτό είναι ένα σημείο ε, αφετηρίας το οποίο πρέπει να το αναλύσουμε. Οι τροποποιήσεις ε, δεν έχουν στόχο μόνο τη διευκόλυνση τη διασυνοριακή συνεργασία σε δεδομένα από αρχές επιβολής του νόμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ε, όχι μόνο από τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και από οποιαδήποτε χώρα σε όλο τον κόσμο, όποια χώρα έχει επικυρώσει τη σύμβαση της Βουδαπέστης ή πρόκειται να το πράξει στο μέλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι πιο συχνές ε, Απόπειρε παραβίαση της εμπιστευτικότητα των ε, ε, εγγράφων προέρχονται από οντότητε που θεωρείται ότι έχουν, μία, έχουν ε, εκ του νόμου τη δυνατότητα πρόσβαση στα εγγράφα αυτά. Κατά την άποψή μα, λοιπόν η επέκταση του πρωτοκόλου σε δεδομένα σε πρόσβαση σε δεδομένα από ιδιωτικέ εταιρείε δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και σοβαρές ανησυχίε σε σχέση με το ποια δεδομένα θα είναι προσπελάσιμα de facto και επί βάσεως. Επίσης και το θέμα των ε, αυθαίρετων αποφάσεων ε, που μπορεί να μην ε, είναι αντικείμενο εποπτείας από ανεξάρτητο φορέα. Επίσης θα διακυβεύεται έτσι το, η αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Πιστεύουμε ότι αυτοί οι κίνδυνοι ισχύουν πολύ περισσότερο λόγω των πρόσφατων προβλημάτων μαζικής ε, ε, πρόσβασης σε δεδομένα. Κάθε φορά λοιπόν που θα χρησιμοποιεί κανείς αυτές τις διόδους συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, ε, που δεν θα μπορεί να αιτιολογηθεί η χρήση αυτών των δεδομένων αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας που όπως, όπως ήδη ισχύει στο πλαίσιο της προστασίας δεδομένων αποτελεί ε, μία παράβαση γιατί δεν στο βαθμό που δεν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Οπότε πρέπει να είστε έτοιμοι για ε, τους κινδύνους αυτών των ε, αλλαγών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να εξετάσουμε το ζήτημα λεπτομερέστερα πριν δώσουμε τη συγκατάθεσή μας επειδή επενδύεται από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς μεγάλη προσπάθεια σε όλη αυτή την ε, συζήτηση, πρέπει να συνεχίσουμε βέβαια ε, με ένα πολύ πιο ενημερωμένο διάλογο. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το εξής. Υπάρχει επίγουσα ανάγκη ε, αλλαγής της σύμβασης της Βουδαπέστης. Ας σκεφτούμε μια περίπτωση που δεν ξέρουμε πού είναι τα δεδομένα και τα δεδομένα αυτά μπορεί ας πούμε να κλαπούν σε μια χώρα που δεν ε, είναι συμβαλόμενο μέρος της σύμβασης. Το, ε, το επιπλέον πρωτόκολλο διαδραματίζει κανέναν ε, ιδιαίτερο ρόλο είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί με νέους, νομι... κανόνες. Έχουμε επίσης τα στοιχεία ότι τρέχουσα πρακτική διασυνοριακής ε, προσ... Ε, πρόσβασης στα γεγονότα βάσει του 32β της σύμβασης ε, δεν λειτουργεί καλά. Η προστασία δεδομένων δεν είναι κάτι που μας απασχολεί που άρχισε τώρα μόλις να μας απασχολεί από το Νοέμβριο του 2011 έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό της, αναγκαιότητας, της αρχής αναγκαιότητας και της ε, αναλογικότητας. Κάτι που φαίνεται στο άρθρο 14 για παράδειγμα που λέει ότι πρέπει να αναλαμβάνεται δράση στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης έρευνας και το άρθρο 15 που βλέπετε τώρα στη διαφάνεια που λέει ότι οι εξουσίες και οι διαδικασίες ε, που προβλέπει η Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες πρέπει να ενσωματώνουν το δικαίωμα της αναλογικότητας. Επομένως η προστασία των δεδομένων δεν είναι μια απέτηση που ε, δεν είναι μια προϋπόθεση που την ε, ανακαλύψαμε σήμερα. δεν είναι εμπόδιο η προστασία των δεδομένων και ούτε δημιουργεί πρόβλημα σε μια ε, επίσημη έρευνα ε, δικαστική ε, στο κυβερνοχώρο που θα εμποδίσει τον εισαγγελέα να διεκπεραιώσει επιτυχώς το έργο του στην περίπτωση ενός ποινικού αδικήματος. Αντιθέτως, στην περίπτωση μιας συγκεκριμένης οποιαδήποτε υποψίας, δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων με το σεβασμό συγκεκριμένων δικλείδων ασφαλείας. Δεν θα τώρα σε πολλέ λεπτομέρειες το δεξιοδικό κατάλογο όλων αυτών των νομικών απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται. Θα τις βρείτε τι πληροφορίες αυτές στην ομιλία μου. Όπως επίσης και για το λόγο για τον οποίο ε, χρειαζόμαστε ε, αυτό το νομικό πλαίσιο. Όλες αυτές οι ε, αμοιβαίες συνθήκες, οι συνθήκες αμοιβαίας νομικής συνδρομής πρέπει να τοποθετούνται σε αυτό το πλαίσιο ποιες συστάσεις τώρα μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Καταρχάς εγώ θα έκανα την εξή σύσταση να ε, μεταφραστεί σε πράξη το δικό σας ψήφισμα και δεύτερον θα ήθελα να εξασφαλίσουμε την άμεση έγκριση της μεταρρύθμισης, ε, του πακέτου μεταρρύθμισης ε, της προστασίας δεδομένων ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο κείμενο ε, στην ε, προστασία των δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου. Στην περίπτωση τώρα ύπαρξη τρίτης χώρας, να σας υπενθυμίσω την εκδοχή του Συμβουλίου για το άρθρο 33 της πρότασης του Συμβουλίου για την ε, οδηγία ε, δικαστικών ε, δραστηριοτήτων. Θα μπορείτε να τη διαβάσετε στην παρουσίασή μου, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Και τώρα όσον αφορά τώρα δεδομένα που προέρχονται από ιδιωτικές εταιρείες σε αρχές επιβολής του νόμου, υπήρξε μία πρόταση από πλευράς Επιτροπής σα για ένα επιπλέον άρθρο 43α όλες αυτές οι δικλείδες ασφαλεία, να, ασφαλείας να λαμβάνονται υπόψη. Δηλαδή άμεση πρόσβαση από διοικητική αρχή από τρίτη χώρα απαγορεύεται εκτός εάν κάποιες ε, εγγυήσεις γίνονται σεβαστές προκαθορισμένες εγγύησεις. Θα ήθελα επίσης να ενθαρρύνω τη βελτίωση. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι δυνατόν να, λειτουργήσει αυτό σε κάθε περίπτωση, αλλά βελτίωση των ε, συνθήκων αμοιβαία ε, νομικής συνδρομής, ε, να είμαστε βέβαιοι ότι λειτουργούν καλά, και να είναι αυτές που διέπουν την άμεση πρόσβαση στα δεδομένα. θα βρείτε συγκεκριμένα λεπτομερή σχόλια σε σχέση με την προστασία των δεδομένων και την πρόσβαση αυτών, ε, ε, τα δεδομένα τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά πρέπει να γίνονται αποδεκτά, να γίνονται σεβαστά ε, σε περίπτωση πρόσβασης από τρίτη χώρα, από τρίτη χώρα. για ποιο λόγο είναι σημαντικό το νομοθετικό πλαίσιο, επίσης το εξήγησα. Το θέμα της εθνικής συγκατάφεσης είναι επίσης πολύ σημαντικό γιατί επικεντρώνεται κανείς ε, στον ε, ενδιαφερόμενο, ε, σε αυτόν που αφορούν τα δεδομένα. Στη σύμβαση υπάρχει μια εντελώς διαφορετική έννοια. Αναφερόμαστε στην οντότητα που έχει την εξουσία να διαθέσει τα δεδομένα. Αλλά ποιος είναι ο ρόλος του, αυτόν του ενδιαφερομένου αυτού που τον αφορούν τα δεδομένα. Τι γίνεται επίσης με την αποτελεσματικότητα μιας ανεξάρτητης εποπτείας, της εφαρμογής της αρχής ε, της σύστασης 87-15 ε, της Επιτροπής. Γι' αυτό ακριβώς ε, συστήνουμε όλα τα συμβαλόμενα μέρη του, της Σύμβασης Βουδαπέστης να προσυπογράψουν και τη Σύμβαση Υπαριθμών 108. Δεν πρέπει να είναι σύμβατα μεταξύ τους αυτά τα δύο πράγματα. Πόσες τρίτες χώρες έχουν πλήρως επικυρώσει την Σύμβαση 108 όμως. Αν μου επιτρέπετε, θα ολοκληρώσω με μία μόνο φράση, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ανεξαρτήτως των πολύ καλών προθέσεων όσων ε, επενδύουν τόσο πολύ ενέργεια για αυτό το θέμα, νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από μια λειτουργική λύση και νομίζω ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι διάφορες επιλογές να είναι ένας δούριος ύπος για την επανεισαγωγή μερικών λύσεων που θέλουμε να παρεμποδίσουμε με τον κανονισμό προστασία δεδομένων. Είμαστε διαθέσιμοι για περαιτέρω συζητήσει, αλλά παρακαλούμε ακολουθήστε και λάβετε υπόψη τις συστάσει ε, που ε, σας κάναμε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπα και στην αρχή ότι υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν βαθύνει πολύ το θέμα τα τελευταία λεπτά, αυτά που είπατε, που αναφερθήκατε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου του Μαρτίου και μετά αναφερθήκατε στα διάφορα στοιχεία, τον κανονισμό και άλλες πτυχές, όλα αυτά έχουν μοιραστεί και θα έλεγα οι νέοι ευρωβουλευτές να τα κοιτάξουν για να καταλάβουν καλύτερα περί τίνος πρόκειται και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν κυρίως αν είσαστε καινούργοι στα θέματα αυτά. Πολύ καλά τα ακούσαμε πριν από λίγο. Αλλά ίσως και για αυτούς που έχουν βαθύνει περισσότερο ενώ τα χρήσιμα. Περνώ λοιπόν τώρα στο τελευταίο τμήμα των παρουσιάσεων. Περνώ λοιπόν στον κύριο Διεδιορόφσκι, ο οποίος είναι Γενικός Επιθεωρητής για την Προστασία Δεδομένων από την Πολωνία και Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και που μου δώσατε επίσης την ε, δυνατότητα να παρουσιάσω τις θέσεις μας για το άρθρο 29, σε σχέση, το άρθρο 29 μάλλον, σχετικά με τις προτινόμενες αλλαγές στη σύμβαση της Βουδαπέστης. Όπως τα γνωρίζετε, η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 όπου συμμετέχουν ε, εποπτικές αρχές από όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πει ότι θέλει απευθείας πρόσβαση των ε, τρίτων ε, χωρών, των ε, αρχών τους δηλαδή επιβολής του νόμου. Σε μια επιστολή, επιστολή η οποία έχει σταλεί στις 5 Δεκεμβρίου του 2013. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι τη θέση μας τη στήριξη η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που ονομάζεται TPD με επιστολή της στις 12 Φεβρουαρίου του 2014. Πολύ σύντομα λοιπόν θα περάσω στις κύριες παρατηρήσεις της θέσης της ομάδας εργασίας, που είναι πολύ κοντά σε αυτά που σας παρουσίασε ο προλαλής σας. Στόχος των τροποποίησεων που προτείνονται στη Σύμβαση είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα δεδομένα των αρχών επιβολής του νόμου. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνει προσέχοντας και και έχοντα υπόψη μας όχι μόνο το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων, αλλά και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εδώ τονίζουμε ότι πριν την σύμβαση του 2001 είχαμε τη σύμβαση 108 για την προστασία δεδομένων που δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ό,τι αλλαγές λοιπόν έχουν να κάνουν με την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι μία από αυτές, πρέπει να συμμορφώνεται σε κάποιες αρχές της αναλογικότητας για παράδειγμα και της αναγκαιότητας. Και επιπλέον όσον αφορά την προστασία των δεδομένων υπάρχουν και άλλες απαιτήσει. Μεταξύ άλλων το θέμα του εφαρμαζόμενου νόμου, της αξίας, όπως και κανόνες που έχουν να κάνουν με την μεταφορά δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός της δικαιοδοσίας των μερών που έχουν υπογράψει την σύμβαση. Όπως θα γνωρίζετε, άλλες χώρες που έχουν επικυρώσει τη σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα δεν συμμετέχουν απαραίτητα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αν λοιπόν εξετάσουμε την πρόταση για την αλλαγή του άρθρου 32 της Σύμβασης της Βουδαπέστης υπάρχουν πέντε προϋποθέσεις, νέες προϋποθέσεις που επιτρέπουν τις αρχές επιβολής του νόμου να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Το δεύτερο και το τρίτο λένε ότι η διασυνοριακή πρόσβαση σε δεδομένα μπορεί να ε, δοθεί χωρίς συνένεση αλλά με νόμιμο τρόπο και καλή την πίστη. Αυτές οι προτάσεις μοιάζουν μεταξύ τους. Ο κύριος, το κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη σαφήνειας. Όλες οι έννοιες αυτές δεν αναφέρονται σε δεσμευτικά νομικά μέσα και δεν διασφαλίζουν ότι οι αρχές κλειδί της προστασίας των δεδομένων θα διασφαλίζονται σε όλες τις χώρες. Το γεγονό δηλαδή ότι δεν υπάρχει ενίος ορισμός με τις διαφορές που υπάρχουν στα νομικά καθεστώτα των μερών που έχουν υπογράψει τη σύμβαση μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την εφαρμογή του νόμου. Και μια που είμαι και νομικός που έχω ασχοληθεί με τα θέματα αυτά από το 2001, από τότε που εγκρίθηκε η σύμβαση, το θέμα της μεταφοράς των κανόνων της σύμβασης για τον κυβερνοχώρο στο εθνικό δίκαιο, είχε να κάνει πολλές φορές με τη μετάφραση των όρων που χρησιμοποιεί η σύμβαση και πώς μεταφράζονται οι όροι αυτοί στην γλώσσα της κάθε χώρας. Κάτι το οποίο έχει δυσκολεύσει συχνά τις χώρες να εφαρμόσουν τις διατάξεις αυτές. Η πρώτη πρόταση τώρα βασίζεται, ή μάλλον θα έλεγα θα έπρεπε να βασίζεται, στην αρχική ιδέα. Ότι δηλαδή εφαρμόζονται αντίστοιχες νομικές βάσεις, το άρθρο 32β, τη σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η σύμφωνη γνώμη για να ισχύσει πρέπει να καλύπτει κάποιες προϋποθέσεις, κάποια κριτήρια. Και ένα, το πιο σημαντικό ίσως εδώ, είναι ότι η σύμφωνη γνώμη πρέπει να έχει δοθεί εκ των προτέρων. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν αρνητικές ε, συνέπειες αν δεν την έχει δώσει το άτομο. Αυτό λοιπόν μπορεί να είναι προβληματικό. Σε αυτό το σημείο βέβαια αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν συχνά παρεξηγήσεις όσον αφορά την έννοια της σύμφωνης γνώμης. Υπάρχουν απόψεις μεταξύ των αντιπροσωπιών που ετοιμάζουν αλλαγές και λένε ότι τη σύμφωνη γνώμη αυτή μπορεί να την δώσουν ποιοι, οι πάροχοι των υπηρεσιών διαδικτύου. Αλλά ένα τέτοιο συμπέρασμα είναι απαράδεκτο από τις αρχές προστασίας δεδομένων. Μια άλλη πτυχή της πρότασης αυτής είναι ότι τα δεδομένα θα μπορούσαν να ε, μεταφέρονται χωρίς περιορισμό σε άλλο μέρος από τα συνυπογράφοντα. Μια τέτοια προσέγγιση όμως, όπως το αντιλαμβάνεται η ομάδα εργασία 29, καλύπτει καταστάσεις όπου είναι ασαφές σε ποια δικαιοδοσία τελικά βρίσκονται τα δεδομένα ή προς τα που μετακινούνται. Η τέταρτη πρόταση εγείρει αντίστοιχε ανησυχίες γιατί επιτρέπει την επέκταση της έρευνας χωρίς περιορισμούς στην επικράτεια της συγκεκριμένης χώρας. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες της εδαφικότητας εδώ, όπως και της κυρίαρχης δικαιοδοσίας μπορεί να παραβιαστούν. Μια προσπάθεια να υπάρξει υποχρέωση για σύμφωνη γνώμη δεν έχει και πολύ νόημα. Η τελευταία πρόταση επικεντρώνεται στο λεγόμενο εξουσία διάθεσης δεδομένων του ατόμου και βασίζεται στην υπόθεση ότι αν δεν υπάρχει γνώση του που βρίσκονται τα δεδομένα θα μπορούσε να επαρκούσε να καθοριστεί που βρίσκεται το άτομο το οποίο ελέγχεται σε σχέση με τα δεδομένα αυτά. Δεν υπάρχει όμως τους ορισμούς των οδηγιών, για παράδειγμα 95-46 ή το πλαίσιο απόφασης 2008-977 εξαρτώνται από το πλαίσιο δραστηριοτήτων και το που είναι εγκατεστημένος ο ελεγκτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί με το που βρίσκονται τα δεδομένα. Όπως βλέπουμε λοιπόν, οι κύριες ανησυχίες εδώ πέρα μοιάζουν μεταξύ τους. Το θέμα του πιο δίκαιο εφαρμόζεται και στη συνέχεια αν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι εκπρόσωποι της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 που συμμετείχαν στις συζητήσεις παρόλο που βοηθήθηκαν όλες οι πλευρές να κατανοήσει καλύτερο ένα τον άλλον παρόλα αυτά η αντιπροσωπεία της ομάδας εργασίας 29 είχε την εντύπωση ότι μάλλον οι συμμετείχοντες δεν κλείνουν στην ε, σωστή ισορροπία μεταξύ όλων των πλευρών. Αλλά χρειάζεται περισσότερη ανάλυση. Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 δουλεύει πάνω σε αυτά και σκοπεύει να παρουσιάσει περισσότερα δεδομένα για να διασφαλιστούν επαρκή επίπεδα προστασίας. Συνεχίζεται η συζήτηση και περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα στην ομάδα εργασίας του άρθρου 29 στα τέλη του Νοεμβρίου. Ένα από τα θέματα της συζήτησης στην τελευταία συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ακριβώ αυτό. Λαμβάνοντα υπόψη λοιπόν τώρα την επιθυμία μα να έχουμε περισσότερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολή του νόμου και λαμβάνοντα υπόψη μα ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο να το κάνουμε, Λαμβάνοντα επίση υπόψη ότι η συμμόρφωση με τι απαιτήσει για την προστασία των δεδομένων διασφαλίζεται με διαφορετικά μέσα, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνε για την προστασία αυτή που να ισχύουν πάντα. Προετοιμάζοντα νομική δράση, κάποιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλο το πλαίσιο, όχι μόνο το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νομοθετικό, αλλά και εκείνο του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο υπήρχε ήδη όταν ετοιμάστηκε η σύμβαση. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί η σύμβαση είναι ανοιχτή για υπογραφές προς τις χώρες που δεν έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την ε, Σύμβαση 108. Γι' αυτό ακριβώς είναι ζωτική σημασίας να έχουμε αρκετές προδιαγραφές προστασίας δεδομένων στην ίδια τη Σύμβαση της Βουδαπέστης. Εμείς στηρίζουμε ότι χωρίς το κατάλληλο πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν πολύ νωρίς να τροποποιήσουμε την σύμβαση έτσι όπως προτείνεται μέχρι τώρα. Και επιπλέον θέλω να υπενθυμίσω και κάποια πράγματα που είπα εδώ στην Επιτροπή σας πριν από δύο χρόνια, που είπαμε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δραστηριότητες προστασίας δεδομένων είναι σύνεκβανομ συνθήκη για να μπορέσει να υπάρξει πραγματική ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής των, του νόμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε που τηρήσατε και το χρόνο σας. Αυτό βοηθάει πολύ. Έχω κατάλογο μιλητών εδώ και θέλω επίσης να σας πω ότι το θέμα αυτό των τροποποίησεων στη σύμβαση της Βουδαπέστης δεν έχει να κάνει μόνο με το ψήφισμα σε σχέση με θέματα ανταλλαγή πληροφοριών, υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά έχει να κάνει και με το ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνας και άλλα θέματα συνεργασίας στον τομέα του εγκλήματος. Έχουμε. Πριν κλείσω τον κατάλογο ομιλητών, κανένας άλλος θέλει το λόγο παρακαλώ. Η κυρία Στίβενς, άλλος κανείς. Κλείνω τον κατάλογο ομιλητών. Σύμφωνη. Καλώς. Η κυρία Σίπολ πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά. Κατά την άποψή μου, τα κρίσιμα σημεία σε αυτή τη μετατροπή της σύμβασης είναι κρίσιμο το θέμα της άμεσης πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων άλλης χώρας. Αν ε, δούμε τα τελευταία πέντε χρόνια τους διάφορους ε, οδηγίες και τις διεθνείς ε, συμφωνίες, πάντοτε ακούγαμε ωραία λόγια ότι όλοι που συμμετέχουν ε, τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, ότι χρησιμοποιούν τα αναλογικά τα δεδομένα, όμως στην πράξη υπήρξε τόσο μεγάλο εύρος χρήσεων που τελικά δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ε, κανέναν. Ε, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι τηρούνται αυτά τα δικαιώματα. Η σύμβαση δεν έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά με τρίτα κράτη που θα προσχωρήσουν στη σύμβαση και αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Από μόνη της η κατάσταση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προβληματική γιατί διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν ενιαία στάνταρ σε επίπεδο προστασίας δεδομένων ούτε και στα νομικά μας συστήματα, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά. Έτσι, λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ε, έχουμε την εμπιστοσύνη ότι θα υπάρχουν ε, συγκρίσιμα στάνταρ στα οποία θα βασιστούμε, πώς γίνεται η αποθήκευση, πώς ε, διεξάγεται η πρόσβαση στα δεδομένα και η μεταφορά τους, η διακίνησή τους. Αν υπάρχει δηλαδή ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλό δε μάλλον στις τρίτες χώρες οι οποίες ε, θέλουν να προσχωρήσουν στη σύμβαση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θεωρώ ότι τουλάχιστον είναι επικίνδυνο ε, να προχωρήσουμε έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχουν ε, απίστευτες συνέπειες αν ακολουθήσουμε την ταχεία οδό και δώσουμε αμέσως πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων άλλων χωρών χωρίς να έχουμε έλεγχο για το τι θα συμβεί με αυτά τα δεδομένα ή ε, έλεγχος για τα νομικά συστήματα, με, ποιες, ε, με ποια τεκμήρια χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα στις νομικές διαδικασίες. Επίσης, πώς συλλέγονται τα δεδομένα. Ε, πολλές ε, φορές ε, αυτό μπορεί να, ισχυ... να γίνεται κάπως ένα εθνικό σύστημα που να μην ισχύει το ίδιο σε κάποιο άλλο. Επίσης, η ποινική δίωξη θέλουμε να πάει πιο γρήγορα, αλλά πάντοτε δεν μπορούμε να το πετύχουμε λόγω των διαφορών. Πώς λοιπόν θεωρούμε ότι έχοντας πρόσβαση στους σερβερ και στα εις δεδομένων άλλων χωρών θα έχουμε ε, λύσει αυτό το πρόβλημα. Εγώ δεν θα συμφωνούσα σε καμία περίπτωση σε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Η Σόφη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμμερίζομαι πλήρως τον σκεπτικισμό που έχει ήδη εκφράσει η κυρία Ζήπολ, γιατί ειλικρινά οι δύο πρώτοι ομιλητές, μην το πάρετε προσωπικά, ε, δεν είναι καθόλου αξιόπιστοι ως προς τα λόγια τους, διότι καταρχάς ε, αντιφάσκεται. Εσείς λέτε, κύριε ε, Πλάγκεν, απρόσκαπτη πρόσβαση όχι, δεν με καταλάβατε καλά και ο επόμενος ομιλητής είπε ότι είναι πολύ καλή ιδέα. Τελικά ποιο από τα δύο ισχύει. Ήμουνα μέλος αυτή της Επιτροπής ε, τα τελευταία δέκα χρόνια και πραγματικά δεν μπορώ να σας πω πόσες φορές μας έχουν ε, βεβαιώσει ότι υπάρχουν νομικές δικλείδες ασφαλείες. Κοιτάξτε, Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ε, θεωρείτε ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε τις κυβερνήσεις. Κύριε Πλάνκεν, εσείς και εγώ τις ξέρουμε πολύ καλά. Αυτές τις κυβερνήσεις ε, που χρησιμοποιούν πρακτικές καουμπόι και κάνουν ε, παράνομες παρεμβάσεις και έχουν παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα. Αν δεν μπορείτε να τα τεκμηριώσετε αυτά, να μην έρχεστε εδώ. Αν ε, οι κυβερνήσει μπορούν από μόνε τους να μπαίνουν στα δεδομένα μας, ε, μην έρχεστε εδώ να μας τα λέτε αυτά και να ζητάτε την υπογραφή μας. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε τις κυβερνήσεις όταν οι Βρετανικές μυστικέ Υπηρεσίες αρνούνται ότι εξ αποστάσεως ενεργοποιούν τις κάμερες ε, και παρεμβαίνουν στην ιδιωτική μας ζωή στα σπίτια μας. Θέλετε να συμπράξουμε, να υπογράψουμε μια τέτοια σύμβαση. Ελάτε τώρα, πραγματικά αν είστε σοβαροί για αυτές τις νομικές διασφαλίσεις, αγαπητοί κύριοι, πηγαίνετε στις εθνικές κυβερνήσεις και πείτε τους να επιταχύνουν την έγκριση του πακέτου προστασίας δεδομένων με μια αποδεκτή μορφή και τότε ξαναμιλάμε, τότε ξαναμιλάμε. Και αυτό είναι το μόνο που είναι αποδεκτό για μένα. Και πραγματικά γίνομαι όλο και πιο κοινική. Δεν πρόκειται να αναλάβω καμία ευθύνη για μία νομιμοποίηση παράνομων πρακτικών. Αυτό είχα μόνο να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στη μάχη κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος το Κοινοβούλιο έχει αφιερώσει πολλή δουλειά. Υπάρχει η οδηγία για αυτό το θέμα, η οδηγία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Πρόσφατα εγκρίναμε το ευρωπαϊκό ένταλμα, την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας ε, που δείχνει ακριβώς ε, πώς ε, για, την εφαρμογή του νόμου πρέπει να υπάρχει συνεργασία εντός της Ευρώπης. Αυτά είναι θέματα για τα οποία έπρεπε να μαχηθούμε έναντι των κυβερνήσεών μας, έτσι ώστε να έχουμε ένα αξιόπιστο και νόμιμο περιβάλλον. Η νομιμότητα λοιπόν αυτών των προτάσεων είναι αμφισβητήσιμη. Καταρχάς να πω και να προτείνω να σταματήσουν οι συζητήσεις στα κράτη-μέλη και στην Κομισιόν αν δεν ξεκαθαριστεί αν υπάρχει νομική βάση για να υπογραφεί αυτή η συνθήκη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δηλαδή, καν να την συζητήσουμε γιατί σε αυτό το θέμα το η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητές της. Δεν... Είναι λοιπόν νόμιμο τα κράτη-μέλη να διαπραγματεύονται εντό του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Άρα η νομική υπηρεσία θα πρέπει να μας δώσει την γνωμοδότησή της για να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο, αν μπορεί να γίνει. Τον Απρίλιο επίση υπήρξε από το ΔΕΚ μια απόφαση για την φύλαξη δεδομένων στο περιβάλλον των επικοινωνιών. Και όπως ε, μπορεί σίγουρα να γνωρίζετε, το δικαστήριο έκρινε την οδηγία 26-24 για την ε, ε, τυφλή φύλαξη των δεδομένων και μίλησαν και για την εδαφικότητα και φαίνεται εκεί ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη της είναι παραβίαση να μεταφέρουν δεδομένα, να διαβιβάζουν δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και όλων των πολιτών στην Ευρώπη σύμφωνα με το άρθρο 7 για την ιδιωτική ζωή και την οικογενειακή ζωή. Επίσης, δεύτερον, Υπάρχει αυτή η έννοια που στην ουσία ε, εναπνεύστη το συνταγματικό δικαστήριο του, της Γερμανίας που μιλάει για την ακεραιότητα και το απόρριτο των συστημάτων πληροφορικής. Η ελεύθερη πρόσβαση σε τέτοια συστήματα θα ήταν ε, κατάφορη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπάρχουν πολύ ψηλά στάνταρτ τα οποία έχουν εναρμοτιστεί εναρμονιστεί μεταξύ των κρατών μελών για αυτή τη σύμβαση. Δεν το βλέπω και ε, δεν το βλέπω γιατί στην ουσία υπάρχει περιορισμός ε, Λόγω της απόφασης του δικαστηρίου υπάρχει η ιδιωτική ζωή. Δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε ένα σύστημα που μπορεί να περιλαμβάνει ας πούμε το ημερολόγιό μου. Αυτό αναφέρεται σε αποφάσεις των δικαστηρίων ε, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτά τα πράγματα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαριστούν. Μετά λέτε ότι ε, δεν υπάρχουν κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Κοιτάξτε, υπάρχει, υπάρχει η οδηγία του 95 ε, που προστατεύει τα δικαιώματα, τα δεδομένα, συγγνώμη. Θα έπρεπε να το ξέρετε αυτό. Και ως προς την ουσία να πω ότι κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία. Το πρωτόκολλο που ε, προτείνεται θα είναι παραβίαση του άρθρου 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και για να καταλήξω να πω ότι είναι καλό που μιλάμε για την αμοιβαία αναγνώριση και για την προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας, γιατί μαθαίνουμε από αυτό, ας πούμε, με το ένταλμα σύλληψης μάθαμε με τον δύσκολο τρόπο ότι δεν είναι καλό να αντικαθιστούμε ένα κενό στον νόμο στην πλευρά της ασφάλειας με ένα άλλο κενό στην πλευρά των θεμελιωδών δικαιωμάτων, πραγματικά δεν είναι σοφό να πράττει κανείς έτσι. Ε, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς εναρμόνιση και πραγματικά αυτή τη στιγμή όλα τα μέρη που θα πρέπει να υπογράψουν τη σύμβαση θα πρέπει να έχουν κοινά στάνταρ και αυτό δεν το έχουμε δει. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται το κείμενο γιατί δεν έχουμε αυτά τα στάνταρ. Τέλος, η θέση μας το Μάρτιο για την, στην έκθεση για τις μαζικές παρακολουθήσεις είχε να κάνει και με το θέμα της δημιουργίας εμπιστοσύνης στη συνεργασία που έχουμε για την πάταξη του διασυνοριακού εγκλήματος. Δεν μπορεί να είναι μονομερής αυτή η εμπιστοσύνη. Χρειαζόμαστε καλύτερη εφαρμογή και εκτέλεση των υφιστάμενων κανόνων που ήδη υπάρχουν δηλαδή στη σύμβαση, να βελτιώσουμε την κατάσταση και να προωθήσουμε και να πιέσουμε για διασφαλίσεις πραγματικά δεν γίνουν αυτά, ε, δεν θα μπορούσα ε, να μιλήσω για περαιτέρω συνεργασία. Η Σύμβαση 108 πρέπει πρώτα να βελτιωθεί, γιατί αυτή είναι η βάση όλων. Ευχαριστώ, Γιάν. Δεν θέλω... Ε, να πω ότι είχα κάποιο λόγο που δεν ανέφερα το, την εντολή, το ευρωπαϊκό ένταλμα διερεύνησης είχα λάβει μέρος σε αυτό. Να πω ότι πραγματικά ε, υπήρξε μεγάλη συνεργασία από όλα από όλες τις ομάδες, τις πολιτικές, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο το οποίο να είναι αξιόλογο και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω ότι έπρεπε να το πω αυτό τώρα στη συζήτηση για τη Σύμβαση της Βουδαπέστης. Επόμενος ομιλητής τώρα η κυρία Μουσολίνη. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, επιτέλους ο μιλητής που πήρε το λόγο ακριβώς πριν από μένα είπε πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία απουσίαζαν από τις παρουσιάσεις των προσκεκλημένων μας. υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δικαιωμάτων. Από τη μία είναι η πρόσβαση στα δικαιώματα και από την άλλη είναι η προστασία των δεδομένων. Και υπάρχει και το θέμα της πληροφορικής. Στην Ιταλία είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες μόνο για αυτούς θα μιλήσω παρά το γεγονός ότι δεν είναι μόνο ε, ευρωπαϊκό ζήτημα. Εμείς εκπονούμε τόσους πολλές ε, ε, συμβάσεις, τόσα πολλά πρωτόκολλα, αλλά δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί καταγγελίας. Το, δεν είναι οι μηχανισμοί από τους με τους οποίους μπορούμε να καταγγείλουμε κάτι. Τα θύματα ενός αδικήματος ε, ε, στον κυβερνοχώρο, πού θα καταγγείλουν το πρόβλημά τους. θα μπορούσε να υπάρχει ένα εικονίδιο στο οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κλικ στον υπολογιστή μας και να έρθουμε σε επαφή με, ένα ε, ε, αστυνομικό, μια αστυνομική υπηρεσία για παράδειγμα, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με άλλους οργανισμούς, ε, με ε, αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλες χώρες. Είναι όμως αυτό πάρα πολύ περίπλοκο. Εμένα με απασχόλησαν αυτά τα θέματα, τα μελέτησα Έχουμε μια καινούρια σύνθεση αυτή τη στιγμή ως Επιτροπή, αλλά ο χρήστης, ε, ο νέος χρήστης του διαδικτύου ε, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα συστήματα πληροφορικής δεν έχει ένα μέσο καταγγελίας. Εντάξει, εγώ δεν λέω να καταγγείλουμε τα αδικήματα αυτά, αλλά σε ποιου, ποιοι είναι οι συνομιλητές μας. Μιλάμε για τη σύμβαση της Βουδαπέστη, αλλά είμαστε σοβαροί. Χρειαζόμαστε ένα απλό αποτελεσματικό μέσο προσπελάσιμο για τις καταγγελίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Και η κυρία Στίβεν, πριν ε, δώσουμε και πάλι το λόγο στου προσκεκλημένους μας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, άκουσα πάρα πολύ καλά όλους τους συναδέρφους. Αυτό το θέμα είναι κάπως καινούριο για μένα. Γι' αυτό είμαι προσεκτική. Υπάρχουν προβλήματα από ό,τι καταλαβαίνω για να πετύχουμε την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του ιδιωτικού βίου και την προστασία των δεδομένων από τη μία και από την άλλη μεριά έχουμε το δικαίωμα των ε, αρχών να μπορούν να βρουν πληροφορίες για να αποφεύγουν εγκληματικές πράξεις. Εδώ όμω υπάρχει και κάτι άλλο. Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει σκάνδαλα όπου οι μυστικές υπηρεσίες εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εμπλεχτεί και καταλήγουμε έτσι σε μια περίεργη κατάσταση γιατί αυτές οι χώρες έχουν συνυπογράψει τη σύμβαση. Ενώ κάνουν παράνομα πράγματα. Άρα τίθενται όντω ερωτήματα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και αν δούμε το απόρριτο, κάποτε ήταν απόλυτο. Τώρα, στους σύγχρονους καιρούς, η προστασία του ιδιωτικού βίου δεν είναι πια τόσο απόρριτο. Οι καιροί αλλάζουν. Πρέπει να αλλάζουμε κι εμείς. Η προστασία όμως του ιδιωτικού βίου είναι κάτι ζωτικής σημασίας. Και όταν πρόκειται για εγκληματικέ πράξεις, πρέπει να ισχύει η αναλογικότητα και να την, προστατεύουμε, κάτι το οποίο λείπει σε αυτά που ακούμε κάπως. Πολλές χώρες έχουν επικυρώσει τη σύμβαση, μάλλον έχουν υπογράψει τη σύμβαση χωρίς να την έχουν επικυρώσει. Παραμένουν 11 χώρες που δεν την έχουν επικυρώσει ακόμα. Η σύμβαση του 2001, έτσι, έχουν περάσει τόσα χρόνια και στο μεταξύ δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση χώρες αυτές. Δεν θα έπρεπε να στείλουμε ένα μήνυμα στις χώρες αυτές, γιατί είναι περίεργο. Στη Ρωσία, για παράδειγμα, τι συμβαίνει. Η Ρωσία είναι εταίρος στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά δεν το έχει κάνει. Πολύ σημαντικός παράγοντας και να μην ε, μιλήσουμε και για την Κίνα, έτσι. Άρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και ελπίζω όλες οι χώρες να συνεργαστούν ώστε να προστατεύονται τα άτομα και ιδιωτικό τους Σε Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Στίβενς. Ε, σας ε, έγιναν ε, έτσι, κάποιες έντονες ερωτήσεις και έντονα σχόλια. Τρία λεπτά να δώσω στον καθένα σας. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να τα καταφέρετε και να απαντήσετε στις ερωτήσεις ε, που σας απευθύνθηκαν και ειδικότερα τις πιο επίμαχες. Να αρχίσουμε και πάλι με τη σειρά των, που έγιναν και οι παρουσιάσεις. Ερικ Πλάνκεν πρώτα. Παρακαλώ, τρία λεπτά, αν μπορείτε. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να ξαναπάρω το λόγο και ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές που μου έθεσαν ε, ερωτήματα. Βλέπω κινησμό, βλέπω έλλειψη εμπιστοσύνης, δυσπιστία, βλέπω ε, και σύγχυση. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. σχόλιο εκτός μικροφώνου που δυστυχώς δεν ακούμε. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι κανόνες ε, του Κοινοβουλίου, αλλά παρακαλώ, απαντήστε, λέει ο Πρόεδρος. Uh, to cynicism, I must say. Στον κινησμό αυτό, απαντώ το εξής. Έχουν γίνει πολλά Όμως έχω την εντύπωση ότι αυτά που λέμε μεταφέρονται κάπως λάθος και και είναι σαν να μου λέτε ότι εμάς ε, μας ε, ε, επηρεάζουν υπηρεσίες μυστικές ενώ εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω εκ μέρους των αρχών ε, επιβολής του νόμου και εξ ονόματος αυτών ζητούμε μια πρόσκοπτη πρόσβαση στα δεδομένα. Δεν θέλουμε απρόσκοπτη όμως πρόταση, ε, συγγνώμη, πρόσβαση για οποιοδήποτε ε, σκοπό. Μιλάμε για ποινικά αδικήματα και μιλάμε για πρόσβαση δικαιολογημένη ε, όταν πρόκειται πάντοτε για εγκληματικές δραστηριότητες. Και νομίζω ότι αυτό το καταστήσαμε σαφές, αλλά δεν ακούσαμε πολλές απαντήσεις σε σχέση με αυτό. Ε, η Επιτροπή Λίμπε θα εξασφαλίσει ότι προστατεύονται τα δικαιώματα των ανθρώπων και οι περιουσίες τους ε, και πώς θα τους προασπίσει, πώς θα τους υπερασπίσει απέναντι στα εγκληματικά, ε, απέναντι στα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και να αποφύγει ένα σενάριο ζούγκλας ή πώς θα αντιδράσει αν το κάθε κράτος μέλος ακολουθήσει τη δική του λύση για τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό νομίζω ότι η Επιτροπή Προστασίας ε, Δεδομένων ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν ε, ένας από τους παραλήπτες της αποστολής της Ομάδας Εργασίας 29 από τα, από τις, από μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είναι ε, μέρη στην ε, Σύμβαση της Βουδαπέστης, μόνο δύο δεν έχουν επικυρώσει. Και επίσης έχουν υπογράψει και τη Σύμβαση 108. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σίγκερ. και εμείς αλλά και άλλοι συνάδελφοι που ε, ασχολούνται με το θέμα αυτό, δεν θα υπά... είπαμε ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία καθόλου ε, όσον αφορά τα ε, εγκλήματα. Εμείς συνεργαζόμαστε με τις διάφορες χώρες για την εφαρμογή της Σύμβασης ε, της Βουδαπέστης αλλά και για την εφαρμογή της Σύμβασης 108 και είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι οι ίδιες χώρες που ασχολούνται με νομοθεσία για τα κυβερνοεγκλήματα ασχολούνται και με την νομοθεσία που αφορά την προστασία των δεδομένων. Αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη. Τώρα, για την ε, αμοιβαία νομική συνδρομή αν δει κανείς ε, τις ε, συζητήσεις ε, του 2012, η πρώτη επιλογή ήταν να είναι πιο αποτελεσματική αυτή η αμοιβαία συνδρομή και η αξιολόγηση που γίνεται από την Επιτροπή που ασχολείται με το έγκλημα του, στον κυβερνοχώρο είναι, ασχολείται με το θέμα της εφαρμογής του άρθρου 31 και Επίσης συζητιούνται οι 20-30 συστάσεις που έχουν προκύψει από αυτήν την ε, Επιτροπή. Να μην ξεχνούμε λοιπόν ότι δεν έχει καμία αιμονή με την πρόσβαση στα δεδομένα αυτή η Επιτροπή. Απλώς είναι ένα από τα, από τα σημεία που την απασχολούν. Όσον αφορά τώρα την ελεύθερη, απρόσκοπτη ε, πρόσβαση, νομίζω ότι ευρωβουλευτής που έθεσε το ερώτημα αυτό, εμείς δεν είπαμε εξ αποστάσεως απρόσκοπτη πρόσβαση στα δεδομένα, ε, δεν είπαμε ποτέ τέτοιο πράγμα. Η σύγχυση μεταξύ της ε, ποινική δικαιοσύνης αλλά και της πρόσβασης είναι ένα θέμα ε, το οποίο Το κάλυψε νομίζω και ο συνάδελφος από την ομάδα εργασίας 29. Ε, Έχει να κάνει και με το πού βρίσκεται ο ε, επόπτης των δεδομένων, πού βρίσκονται τα δεδομένα. Ε, είναι και το θέμα της, αυτό μας φέρνει και πάλι στο θέμα της εξουσίας για τη διάθεση των δεδομένων. Αν δεν ξέρει κανείς πού είναι τα δεδομένα, αλλά είναι εδώ ο ενδιαφερόμενος που τον αφορούν τα δεδομένα, γιατί να μην χρησιμοποιήσω, να μην ακολουθήσω τους κανόνες ε, της, ε, της δικής μου χώρας. Ε, αυτό εννοούσαμε ως προς την εξουσία διάθεσης των δεδομένων. Και αυτό που είπε ε, επίσης ο εκπρόσωπος από την ομάδα εργασίας 29 για τη συγκατάθεση ναι, το τονίσαμε αυτό και είναι κρίμα που η επιστολή αυτή του Δεκεμβρίου δεν έλαβε υπόψη ε, τις ε, τελευταίες ε, εξελίξεις του Νοεμβρίου και ουσιαστικά η επιστολή κάλυπτε προηγούμενη εκδοχή του κειμένου. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να επαναλαμβάνουμε διαδικασίες που έχουμε συμφωνήσει. Το θέμα είναι να συνεχίσει η συζήτησή μας. Και το τελευταίο ερώτημα που θα ήθελα το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να πω προς τον κύριο Μπουταρέλη νομίζω είναι ότι πάρα πολύ καλά μας είπατε ε, πώς μπορούμε να ε, εντοπίσουμε τις λύσεις, πώς είναι δυνατόν να εντοπίσουμε λύσεις ή δικλείδες ασφαλείας εάν η Επιτροπή Λίμπε διαφωνεί με, με, την, ε, με το οποιοδήποτε πρωτόκολλο. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Γιάν, έχεις ένα διαδικαστικό? Ναι. Απλώς θα ήθελα για τα πρακτικά να πω ότι είναι κάπως προσβλητικό το να λέτε ότι δεν μας ενδιαφέρει η καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος πέντε χρόνια ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Προσπαθήσαμε να ε, δημιουργήσουμε ένα κέντρο ε, ε, έρευνας των κυβερνοεγκλημάτων που προσπαθεί πραγματικά να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα και βλέπουμε ότι η δουλειά αυτή δεν συνεχίζεται, αλλά αρχίζουμε μια άλλη διαδικασία που θεωρούμε ότι δεν παρέχει καμία εγγύηση ε, και πραγματικά νομίζω ότι αυτό είναι προσβλητικό γιατί είπατε κιόλας ότι δεν θα υπήρξε καμία ε, συνεργασία σε ποινικά θέματα αν ακολουθήσουμε αυτά που λέγονται εδώ από την Επιτροπή μας. Όχι, πραγματικά αυτό είναι σαν να ε, υποτιμάτε τον ίδιο σας τον εαυτό. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία, υπάρχει αμοιβαία συνδρομή. Λαμβάνει χώρα η συνεργασία αυτή, διμερώς μεταξύ των κρατών μελών και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το αγνοήσετε αυτό και είπατε ότι δεν συμβαίνει αυτό, προφανώ καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται κάτι καινούριο. Ναι, και εγώ στο ίδιο συμπέρασμα θα κατέληγα, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, αυτό δεν ήταν διαδικαστικό, Γιάνν παρά το γεγονός ότι εγώ είμαι ο πρόεδρος της Επιτροπής, είναι αλήθεια ότι έχουμε ένα ε, όγκο εργασίας, ε, το οποίο φαντάζομαι το γνωρίζετε κι εσείς κύριε Πλάνκεν, εσείς μιλήσατε για αυτό το θέμα του σεναρίου της ζούγκλας, το καταλαβαίνω αυτό που είπατε, αλλά και εμείς έχουμε πάρα πολύ δουλειά πίσω μας για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυφέρνο χώρο. Ε, έχουμε πάρα πολύ νομολογία υπόψη μας και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ ε, για τον τομέα αυτό. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι διαδικαστικό, ε, είναι κάτι το οποίο έπρεπε να ακουστεί και αυτό. Τώρα, κοιτάξτε, δεν θέλω να πείτε σε διάλογο, γιατί προφανώς υπάρχει διάσταση απόψεων, οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω το εξής να ακούσουμε και τα υπόλοιπα σχόλια, το τέλος της παρουσίασής σας και κάποια συμπεράσματα, αλλά δεν με πειράζει να γίνονται ζωηρές συζητήσεις, ε, Μπορεί κάποιοι ευρωβουλευτές ε, να μην γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι η σύμβαση της Βουδαπέστης και γιατί γίνεται αυτή η ζωηρή συζήτηση. Είναι γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή τη σύμβαση μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό ακριβώς καλώς είναι πάρα πολύ ε, ε, έντονη συζήτηση. Λοιπόν, ο κύριος Μπουταρέλη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνυπογράφω όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι σήμερα. και οι ευρωβουλευτές και η κυρία Βέλτ και η κυρία Σέγγελ και ο Γιάνν Άλμπερτ. Μερικές φορές και εγώ προσπαθώ έτσι την ορμή μου να τη συγκρατώ, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Έχουμε, οπότε το καταλαβαίνω. Και είμαι και γνώμων στην κυρία Μουσολίνη, η οποία ανέφερε κάτι πολύ βασικό, τα θύματα. Πώς δηλαδή να καταγγέλουν τα θύματα τις εγκληματικές δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο. Όντως, πρέπει να ακούγεται η άποψη των θυμάτων. Επιμένω όμως και στο προηγούμενο συμπέρασμά μου. Και δεν θέλω εδώ να με παρεξηγήσετε, γιατί όταν λέω ότι ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί μεταξύ ειδικών, δεν εννοώ ότι έχουμε τη βάση για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, γιατί το σχέδιο κανονισμού οδηγίας, οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, έχουν πρόβλημα να συνεχίσουν τη συζήτηση για λύσεις οι οποίες αντιβαίνουν στο άρθρο 53α του σχεδίου που λέει ότι όταν έρχεται έτοιμα από μια διοικητική αρχή άλλης χώρας, τότε ο ελεγκτής πρέπει να κοινοποιήσει πρώτα στις αρχές προστασίας δεδομένων και συνεπώς δεν λαμβάνεται απόφαση από άλλη διοικητική αρχή, κυρίως από τρίτη χώρα, δεν προχωράει αν δεν έχει δίπλο ελεγχθεί προηγουμένως. Αν λοιπόν πάμε πίσω στις εναλλακτικέ λύσεις που συζητάμε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι το άρθρο 32β της Σύμβασης ήδη επιτρέπει την άμεση πρόσβαση. Και αυτό είναι ο κίνδυνος για τη σημερινή συζήτηση η αρχή επιβολή των νόμων σήμερα μπορεί χωρίς να ζητήσει τη γνώμη των αρμοδίων ε, αρχών να έχει πρόσβαση στα δεδομένα αρκεί να έχει την συνένεση για τη διάθεση των δεδομένων. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και μετά για να λυθούν κάποια προβλήματα όσον αφορά δυσκολίες εντοπισμού της τοποθεσίας όπου βρίσκονται τα δεδομένα ή εντοπισμού του ιδιοκτήτη των δεδομένων, συζητάμε πέντε δυνατότητες, οι οποίες είναι ζωτική σημασίας. Θα έπρεπε, αντί να παρακάψουμε τη συνένεση, να δίνουμε την δυνατότητα στα τρίτη μέρη να έχουν πρόσβαση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη μας την εδαφικότητα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, πώς να το πω, δεν μας βγάζει πουθενά. Διευκολύνοντας τις έρευνες, βοηθάμε και υπάρχουν προγράμματα, αλλά η σύγκρουση είναι τόσο προφανής και δημιουργεί προβλήματα στο διάλογο και γι' αυτό δεν προχωράμε. Ευχαριστούμε κύριε Βουτερέλη, Ο κύριος Βιερολόσκι. Ευχαριστώ. Τρία σημεία θέλω να θίξω. Πρώτον, είναι αλήθεια ότι υπάρχει παρεξήγηση όταν μιλάμε για την εθνική ασφάλεια και την δικαιοσύνη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. βλέπουμε ότι όλα θα συμπεριληφθούν στην ε, δικαιοσύνη κατά τον κλίματος. Από αυτό που είπε ο Τζοβάνη στην παρουσίασή του, η σύμβαση δεν έχει να κάνει μόνο με την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, αλλά και με τη συλλογή δεδομένων για οποιοδήποτε έγκλημα. Είναι ευρύτερο δηλαδή. Όσον αφορά τώρα τις αρχές επιβολής του νόμου, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποιο είναι το τοπίο των υπηρεσιών αυτών επιβολής του νόμου στις διάφορες χώρες. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πέρυσι το διαπιστώσατε ακόμα και στις ευρωπαϊκές χώρες που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε ποιες είναι οι αρχές επιβολής νόμου διαπιστώνουμε ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχει εποπτεία ή όχι σε αυτές. Γι' αυτό να θυμόμαστε ότι ο κατάλογος των χωρών που είναι μέρη της Σύμβασης για την Καταπολέμηση του Κυβερνοχώρου είναι πολύ ευρύτερος από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν πολλές χώρες εκτός του Συμβολίου της Ευρώπης που συμμετέχουν σε αυτήν. Αυστραλία, άρα η Αυστραλία να μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα, Αμερική, Αζερβαϊτζάν. λέμε να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που είναι σε άλλες χώρες. Τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν επικυρώσει ακόμα την σύμβαση για το έγκλημα. Σε κάποιες από αυτές όμως η διαδικασία επικύρωσης συνεχίζεται. Στο όνομα της ομάδας λοιπόν του άρθρου 29 σας λέω ότι θα συνεχίσουμε στην πράξη το έργο μας με εκπροσώπους από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Γιατί πολύ πρακτικά μπορεί κάποια πράγματα να αλλάζουν από μήνα σε μήνα. Μπορεί να έχουμε πάλι την συμφωνία του SP. Άρα η συζήτηση συνεχίζεται. Συγχρόνως είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία πρακτικά. Παρόλο που, παραλαμβάνω, η συζήτηση καθ' άλλο είναι. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ όλους τους καλεσμένους και ομιλητές μας. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές τη σημασία που έχει αυτό το θέμα. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα μπροστά μας, την νομική συνδρομή, την αναγνώριση, την προστασία του ιδιωτικού βίου, όλα αυτά είναι θέματα που θα έρθουν και θα ξανάρθουν όταν συζητάμε για την εποπτεία και τον έλεγχο. Και πρέπει να το έχετε υπόψη σας. Θα μας απασχολήσουν συνεχώς όταν συζητάμε για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και την προστασία του ιδιωτικού βίου. Σας ευχαριστούμε πολύ.